αξίωμα του Ευρωβουλευτή. Οι αρμόδιες ε, πολωνικές αρχές με ζήτησαν να άρω την ε, ασυλία του κυρίου Τζάτσεκ Κούρσκ σύμφωνα με το άρθρο 6 παραγραφός 2 του κανονισμού. Το αίτημα αυτό ε, απεστάλησε στην Αρμόδια Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Σας υποθυμερώσω ότι σύμφωνα με το άρθρο 3